I bring the meeting to order, I... Παρακαλώ. Can I start with chairman's announcements first? Λοιπόν, πρώτα ανακοινώ του Προέδρου να καλωσορίσω μία ομάδα επισκεπτών από την ε, εκλογική περιφέρεια της Γκεζίνε Μάισεν γύρω στην, ε, στο Ανόβερο αλλά υπάρχει και κάποιος που είναι από το Έμπτεν και σηκώθηκε πολύ νωρίς για να πάρει το λεωφορείο από το Ανόβερο. Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά. Ελπίζω η επίσκεψή σας να σας διαφωτίσει και ελπίζω να αποκομίσετε καλές εντυπώσεις. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και ελπίζουμε να περάσετε καλά. Δεύτερη ανακοίνωση ε, παρακαλώ επιτρέψτε μου ως πρόεδρος να πω κάτι παραπάνω. Είναι τελευταία μέρα που θα είναι μαζί μου η συνεργάτης μου, η βοηθός μου, η Τζούλια Λαμ, η οποία θα ε, πάρει τώρα μία θέση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μεταφοράς ε, Εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων. Με βοήθησε κατά την πενταετία που ήμουν πρόεδρος και ξέρω ότι και η γραμματεία είναι πολύ ευχαριστημένη και θα ήθελε και εκείνη να εκφράσει τις ευχαριστίες της Τζούλια για την εργασία της. Καλή τύχη, καλή δουλειά Τζούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σου στο παρελθόν. Η συνεδρίαση των συντονιστών στις 20 Φεβρουαρίου και στις 17 Μαρτίου. Στις 20 Φεβρουαρίου λοιπόν έγραψα στην ε, και του ζήτησα να ε, συμπεριλάβουν τα σχόλια των Πρασίνων για την μετάβαση προς ε, τους, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και επίσης έγραψα και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Για την Επιτροπολογία σημειώσαμε το ενημερωτικό δελτίο της 6ης ε, και της 17ης και για τα διάφορα οι συντονιστές είπαν ότι θα επανέλθουν στην ε, παραγγελία νέων μελετών επιπτώσεων και κατά την ε, χθεσινή συνεδρία των συντονιστών δεν κάναμε καμία κατανομή εκθέσεων. Ε, θεωρούμε ότι όσες μένουν πρέπει να κατανεμηθούν, να αποδοθούν δηλαδή σε εισηγητές από το επόμενο κοινοβούλιο. Οι συντονιστές προτείνουν να εγκρίνουμε τις διορθώσεις για της ε, την πρόσβαση στη διεθνή αγορά των λεωφορείων και πούλμαν για τις μελέτες από τα διάφορα θεματικά τμήματα, θεματικούς τομείς πολιτικής. Έχουμε κάποιες πιστώσεις. Ο Νίλς είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Ήθελε να κάνει κάτι για το καλοκαίρι. Του ζητήσαμε λοιπόν να αναλάβει τρεις μελέτες πώς θα περάσουμε από το τρένα στο δρόμο και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε ε, με ε, ε, πολυμεσικούς τρόπους τα λιμάνια. Και επίσης, δεύτερη μελέτη, το κόστος της μη Ευρώπης για τις μεταφορές. Ήταν μια εισαγωγική έκθεση που την έλαβαν ήδη οι συντονιστές για την επιτροπολογία. Σημειώσαμε τα τελευταία ενημερωτικά δελτία και για τα διάφορα. Συζητήσαμε ένα θέμα που έθιξαν οι πράσινοι για το τούνελ μεταξύ Λιών και Τουρίνου, τη χρηματοδότηση και τη διαφάνειά του. Και υπήρξε συμφωνία ότι εγώ θα γράψω στον Επίτροπο Κάλλας να ζητήσω διευκρινήσεις για το πρόγραμμα αυτού του τούνελ, αυτή τη σύραγγα μεταξύ Λιών και Τουρίνου και υπάρχει και μια προφορική ερώτηση για το θέμα αυτό, επενθυμίζω, που έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου. Θα γράψω λοιπόν για το θέμα αυτό στον Επίτροπο. Αυτά από τους συντονιστές υπάρχουν ερωτήσεις από αυτόν. Όχι. Ωραία. Να περάσουμε τότε στις ψηφοφορίες. Σας υπενθυμίζω ότι στις 11 σήμερα θα έρθει ο Αντιπρόεδρος Κάλας για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο Συμβούλιο Μεταφορών. Στις 11 λοιπόν. Αυτά λοιπόν από πλευρά συντονιστών. Ωραία. Είναι σαφή τα πράγματα. Για να κάνουμε μια ψηφοφορία ελέγχου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ωραία λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Να σας υπενθυμίσω για τους νέους κανόνες, να σας υπενθυμίσω τους νέους κανόνες. Η τελική ψηφοφορία είναι ονομαστική πάντα. Επειδή έχουν αλλάξει οι κανόνες του Κοινοβουλίου, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Το μηχάνημα θα, ε, σας, ε, θα καταγράψει την ψήφο σας. Λοιπόν, ωραία. Ποια είναι η πρώτη έκθεση που θα ψηφίσουμε. Έγκριση τη συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για μια πρόταση οδηγίας για τον εξοπλισμό των πλοίων και την κατάρριση της οδηγίας 96-98 Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η συγητής Ντομινίκ Ρικέ μία ψηφοφορία, κατευθείαν λοιπόν ψηφίζουμε, ονομαστική τελική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 32 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια Ντομινίκ και όλοι οι συνεργάτες που εργάστηκαν για αυτό. Επόμενο, συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την πρόταση κανονισμού για την πολιετή χρηματοδότηση της ε, εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά την μόλυνση που προκαλείται από τα πλοία και την θαλάσσια απόλυνση που προκύπτει από τις εγκαταστάσεις ε, αερίου και ε, πετρελαίου. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 30 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον Keith Taylor. Τρίτη ψηφοφορία. Πρόταση κανονισμού. Έγκριση συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τον τροποποιητικό κανονισμό 718 για την ε, ε, πολιτική ρύθμιση μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικού στόλου ε, στις εσωτερικές γραμμές Ναϊάδες άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 υπέρ, 2 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε την Καρίν και τους δικούς της συνεργάτες. Αλλά η επόμενη ψηφοφορία δεν θα είναι τόσο απλή ως αυτές οι τρεις. Επόμενη ψηφοφορία, σχέδιο έκθεσης για την πρόσβαση οδηγίας που καθορίζει τους κανόνες για ορισμένα οδικά οχήματα τις μέγιστες διαστάσεις για το εθνικό και για τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και τα μέγιστα βάρη. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Παρακαλώ ε, μετακινηθείτε λίγο προς τα εκεί για να βλέπω καλύτερα το ΕΛΚ. Δεν θα ήθελα τόσο πολύ να τους βλέπω, αλλά ο Ματιέ θα είχε αντίρρηση αν δεν του έβλεπα καλά. Τροπολογία 49 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκατέσσερα και 133 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, 132 είναι προστίκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 172. Εντάξει, παρακολουθείτε όλοι υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Το ECR έχει μία ψήφο περισσότερη. Παραπάνω. Vote is closed. Πέρασε. 15 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και αυτήν άρχεται η ψηφοφορία για την 171. Ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και αυτήν νομίζω ότι είναι ίδιος ο σχετισμός αλλά άρχεται για την 182 η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι <clears throat> πέρας απορρίπτεται 175-181 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Θέλετε να ελέγξουμε. Καλά. Ωραία να ελέγξουμε την 181. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαεννέα. Μαζί 21, 27, 31, 3, 41 και 8. Όλες μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές να τις ελέγξουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 282. 202 συγγνώμη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κατόπιν. 221 και 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 2.26 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 2.26 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. 2.22.38 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.22 υπέρ απορρίπτεται οπότε και επόμενες τρεις συμβαστική τέσσερα υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. I'm getting there. I'm getting there. They're all different page numbers. Είναι διαφορετική συνειδητοποίηση. 2.37 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 2.37 νομίζω ότι εγκρίνεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 2.39 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 2.39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 Άρχεται. 3.28. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Μα ήμουν σίγουρος. 3.30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.29. Α, καταπίπτει. 3.31 είναι απάλληψη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.38 και 3.39 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε τις 3.38 και 9. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνονται. 3.45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.42 και 3.44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 3.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 346 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Εγκρίνεται. 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 1. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 56 παρακαλώ άρχεται νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά πέρας εγκρίνεται 57 57 που συνδυάζεται με την 56 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 58 με τις ίδιες συνθήκες υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και αυτήν άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε τη 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 69 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρασε απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 'Άρχεται ο έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 70 καταπίπτει. 71 καταπίπτει. Πάντα έρχεται το τσάι την ώρα που ψηφίζουμε. Λοιπόν, 72. Μπένιον, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 112 άρχεται νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορώ να βάλω το σακουλάκι με το τσάι με στο νερό πέρας εγκρίνεται συγγνώμη απορρίπτεται εννοούσα, απορρίπτεται εννοούσα. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 9 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 που μπορεί να συνδυαστεί υπέρ, κατά, αποχές, για να ελέγξουμε, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε τον 125 παρακαλώ άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε τον 127 άρχεται πέρας απορρίπτεται 128 δεν είναι αποδεκτή τελική ψηφοφορία η οποία και άρχεται Είναι όπως ξέρετε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία. Καταγράφονται τα ονόματα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα τώρα. Πριν αρχίσετε να χειροκροτείτε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 35 υπέρ 4 κατά δύο εποχές. Εγκρίνεται. Τώρα μπορείτε να χειροκροτήσετε ή να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε. Συγχαίρω τον εισηγητή. Lightfried. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε συνάδελφοι, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Ήθελα να αναφέρω ότι θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης αλλά και όλους που έδειξαν ε, συμβαστικό πνεύμα αλλά και εκείνους που δεν επέδειξαν συμβαστικό πνεύμα διότι η πρόταση που μας έκανε η Κομισιόν ε, ήταν ε, σε μεγάλη συγχύση αλλά καταφέραμε με σκληρή εργασία να καταλήξουμε σε μία λύση ήταν δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Λάιχτφριντ. Και τους κοιόδης ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας. Λοιπόν, για να δούμε εάν έχουμε εδώ την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το ε, πρόγραμμα ομολόγων έργου. Λοιπόν, ωραία είναι παρόντες οι εισηγητές από την ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Μισό λεπτό για να ε, εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται. Παρακαλώ, περιμένετε. Okay, colleagues, if still got interviews to do, could I... Συνάδελφοι, με όλο το σεβασμό παρακαλώ να αποχωρήσετε αν πρέπει να συνεχίσετε τις ε, συζητήσεις σας ε, ή τις συνεντεύξεις σας γιατί οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την πρωτοβουλία για την έκθεση ομολόγων έργων 2020 ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ενδιάμεση έκθεση για την εξολόγηση προόδου του πιλωτικού σταδίου ε, της Πρωτοβουλίας για την Έκθεση Ομολόγων Έργων 2020, στις 11 Φεβρουαρίου οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕΠ να παρουσιάσουν την έκθεση στην Επιτροπή Μεταφορών. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Δύο μιλητές έχουμε, τον κύριο Κασόνη που είναι επικεφαλής ε, του τμήματος για τη Γερατόμ και τις ε, κλιματικές ε, αλλαγές. Ε, καλά, έχετε ένα τόσο τεράστιο τίτλο που δεν ξέρω πώς χωράει την πόρτα σας. Και ο Κόναντ Μέφη που είναι επικεφαλής των ειδικών συναλλαγών του τμήματος υποδομών της ΕΤΕΠ. 15 λεπτά έκαστος θα έλεγα. Ποιος θα πάρει πρώτος το λόγο, έχετε αποφασίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότι η Ιρλανδία κέρδισε το τουρνουά των έξι εθνών, ναι, παρόλα αυτά παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστούμε που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕΠ σαν αυτή την παρουσίαση. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχει καταλητικό ρόλο στην προώθηση τη πρωτοβουλίας για την έκδοση ομολόγων έργων. Ζητώ συγγνώμη ε, γιατί χάνω τη φωνή μου. Θα δώσω το λόγο στην ΕΤΕΠ αν τυχόν σβήσει τελείως ε, τη διάρκεια της παρουσίασης. Από πλευράς Επιτροπής ε, θα έλεγα ότι τα ομόλογα έργα εντάσσονται σε μια γενικότερη απόκριση πολιτικής ως προς τις νέες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ευρώπης, όπου ο τομέας των μεταφορών είναι κατά πάσα πιθανότητα ένας βασικός ε, τομέας όπου εντοπίζουμε κενά χρηματοδότηση τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Ε, το γενικότερο πλαίσιο πολιτικής ε, πρώτα απ' όλα. Πριν από ένα χρόνο θα θυμάστε ότι εκδώσαμε πράσινη βίβλο για την μακροχρόνια χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και στις 26 Μαρτίου θα εκδώσουμε σχέδιο δράσης ε, για την παρακολούθηση της πρώτης πρωτοβουλίας για διάφορους τομείς όπου θεωρούμε πως συντρέχει ανάγκη να ε, αναβαθμίσουμε την ευρωπαϊκή δράση, ε, μεταξύ των οποίων η υποδομή και η στήριξη της δράσης των μικρομεσαίων. Εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις. Εμείς, ε, το Κοινοβούλιο συγγνώμη, ενέκρινε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και το Συμβούλιο συνέστησε ομάδα εργασίας που σε συνεργασία με την ομάδα υψηλού επίπεδου θα υποβάλει αναφορά τον Νοέμβρη. Υπάρχει και μια γενικότερη συζήτηση σε διεθνέ επίπεδο. Υπάρχει σε επίπεδο G20 ομάδα εργασίας. Ε, τώρα συσκέπτονται μάλιστα στην Αυστραλία όπου συζητούν μεταξύ άλλων το πόσο θα προσελκύσουν επενδύσεις και χρηματοδότηση από τις ε, κεφαλαιογορές ε, για την χρηματοδότηση των αναγκών στις υποδομές. Είναι βασικό ζήτημα σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρα από τον νέο κανονισμό και ως απόκριση μετά την χρηματοπιστωτική κρίση χρειαζόμαστε νέες προοπτικές για ένα θεμελιώδη πυλώνα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ευρωπαϊκής οικονομίας. Χρειαζόμαστε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο παιχνίδι. Ε, μιλάμε για θεσμικούς επενδυτές, ε, ειδικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες ε, και παρεμφερείς φορείς. Θα ήθελα να διατρέξω εντάχει αυτή την ε, ε, διαφάνεια. Ξέρετε ότι έχουμε σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο και άρα υπάρχει ε, με καλύτερη ανάγκη να προσελκύσουμε διεθνή δανειακά κεφάλαια και γι' αυτό χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων αυτό το εργαλείο της πρωτοβουλίας έκδοσης ομολόγων έργων. Βλέπετε σε, αυτό το, σε αυτή τη γραφιστική παράσταση ότι θα πάρουμε και τα στοιχεία για το 2013 σε λίγες μέρες, ε, αλλά προς το παρόν μπορείτε να δείτε ότι το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης υποδομής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά το 2013 κατά πάσα... Το 2013 βλέπουμε να αρχίζει μια σημαντική ε, αύξηση, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σοβαρές ανάγκες ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ΔΕΔ μεταφορών και ενέργειας συγκεκριμένα. Για την αγορά ομολόγων και για την χρηματοδότηση έργων ε, μέσα από αυτά τα ομόλογα έργων, βλέπετε ότι εξέλιψαν τέτοιες συναλλαγές από το 2007 έως το 2012 διότι ε, εξαφανίστηκαν οι μονογραμμικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, τι ήταν αυτές, παρήχαν εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Ε, προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό που δημιουργήθηκε μετά την πάυση της δραστηριότητάς τους με αυτή την πρωτοβουλία έκδοσης ομολόγων. Ε, δεν ξέρω αν είστε εξοικειωμένοι με την αρχή. Ε, η ΕΤΕΠ Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν γίνεται έκδοση ομολόγου από μια εταιρεία ομολόγου δίνει δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ε, από τον προϋπολογισμό ε, της ΕΤΕΠ όταν ε, ε, κατασκευάζεται το χαρτοφυλάκιο. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουμε τον πρώτο κίνδυνο σε περίπτωση ζημιών και η ΕΤΕΠ τον υπόλοιπο κίνδυνο. Η ΕΤΕΠ θα σας εξηγήσει σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ήδη αυτή η αρχή χρηματοδότησης και επίκυνται τις επόμενες ημέρες και νέες συμφωνίες. Ποιο είναι το όφελος. Χάρη σε αυτό το σύστημα ε, καθίστε δυνατή η υλοποίηση προγραμμάτων που αλλιώς δεν θα χρηματοδοτούσαν οι επενδυτές. Επίσης ε, μειώνεται η συνολική τιμή του, ε, αγοραία τιμή του χρηματοδοτικού ε, πακέτου που είναι προς όφελος φυσικά της αναθέτουσας αρχής. Ε, εξαμηνία έκθεση θα υποβάλουμε προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενδιάμεση έκθεση το Δεκέμβρη και πλήρης ε, αναθεώρηση θα ε, ε, κάνουμε το 2015. Το 2016 θα αναπτυχθεί πλήρως η πρωτοβουλία έτσι, ομολόγων. Προτού περάσουμε στην ΕΤΕΠ, να σας πω ότι στον ενεργειακό τομέα ε, δύο συναλλαγές ολοκληρώθηκαν και δύο θα κλείσουν σύντομα από χρηματοδοτική άποψης ε, στον τομέα των μεταφορών. Όλες οι αγορές ε, καλωσόρισαν την πρωτοβουλία ως θετική από πλευράς Επιτροπής και ΤΕΠ, η αγορά των ομολόγων έργων έχει αναζωογονηθεί ε, μετά από την σχεδόν εξαφάνισή της, όπως σας είπα νωρίτερα. Ε, το ΣΕΦ, ξέρετε, το, τη χρηματοδοτική διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, ε, εντάσσεται λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία στο ΣΕΦ έως το 10% του προϋπολογισμού της, του συνδέοντας την Ευρώπη μπορεί να διοχετευτεί στα χρηματοδοτικά όργανα, όπως προβλέπεται και στο σχετικό κανονισμό, το 2012 Ο προϋπολογισμός ήταν 230 εκατομμύρια, μοιράστηκε στι μεταφορέ, ενέργεια και τα ευρυζωνικά και για το 2013-2015 προβλέπεται παρόμοιο προπολογισμό. Η πλήρη ανάπτυξη τη πρωτοβουλία, όπω προείπα, θα αποφασιστεί μετά το 2015 ε, μετά την υποβολή της αξιολόγησης τώρα σχεδιάζουμε σε συνεργασία με την ΕΤΕΠΕ τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία πάλι στα πλαίσια της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη ε, προετοιμάζουμε παραδείγματο χάρη τα δάνεια μειωμένη εξασφάλιση, εγκυοδοσία για προγράμματα μεταφορών όπως συνέβη ε, στον προηγούμενο κανονισμό ΔΕΔ και στο μέλλον ίσως ε, εξετάσουμε και το ενδεχόμενο δημιουργίας εργαλείων ε, ε, χρεογράφων βάσει στοιχείων ενεργητικού των εταιριών. Θα δώσω το λόγο τώρα στην ΕΤΕΠ για να συνεχίσει την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ. Σας ακούσουμε τώρα τον κύριο Μέρφη μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά που κάναμε και ας κάνουμε και κάποια εισαγωγικά σχόλια σε σχέση με αυτά που μόλις ακούσαμε από τον κύριο Κασόνη. Πρώτα απ' όλα ε, αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο για τους επενδυτές που επενδύουν σε προγράμματα. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως ότι η εμπλοκή της ΕΤΕΠ ε, σε αυτό το πρόγραμμα, διότι ως προς τη χρηματοδότηση υποδομών έχουμε μεγάλη εμπειρία και ε, παρέχουμε ποιότητα στους επενδυτές και γι' αυτό την χάνει θετικής υποδοχής από πλευράς των επενδυτών σχόλιο εκτός μικροφώνου. Δεν ακούμε δυστυχώς. Ε, ο στόχος της πρωτοβουλίας ε, είναι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν ε, το ρόλο του τραπεζικού τομέα ε, και βασική κινητήριο δύναμη δεν είναι μόνο η δυνατότητα μακροχρόνιας χρηματοδότηση αλλά και η διαθεσιμότητα αυτής της χρηματοδότησης σε ανταγωνιστική βάση ούτως ώστε οι δημόσιες αρχές να έχουν ε, καλή επιστροφή των επενδύσεων που κάνουν. Ε, ξαναλέω είχαμε θετικές εμπειρίες και θα αναφερθώ σε περιπτώσει, περιπτώσεις, μεμονωμένα έργα. Εγώ τρέχω τις διαφάνειες. Ε, το πρώτο πρόγραμμα ε, ήταν το πρόγραμμα Κάστορ, ενεργειακό πρόγραμμα, 1,4 δις ε, έκδοση ομολόγων ε, ήταν βασικός επενδυτής Anchor Investment, 300 ε, εκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕΠ ε, και προσελκύσαμε επενδυτές, 29 το ρυθμό από όλη την Ευρώπη. Οι συναλλαγές έγιναν στο χρηματιστήριο, 20 χρόνια είναι η χρηματοδότηση και η χρηματοοικονομική όρη ήταν ιδιαίτερα ελκυστική, δηλαδή σε σχέση με ε, τα δημόσια ομόλογα είχαμε 100 μονάδες βάσης ε, παραπάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, σε σχέση με την κατάσταση στην Ισπανία, σε σχέση με τις ανάγκες μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και σε σχέση με τη φύση του προγράμματος και των ομολόγων. Είχαμε και μία δεύτερη έκδοση ομολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο τέλη Νοεμβρίου Επίσης είχαμε καλά αποτελέσματα ως προς το ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές. Τρεις φορές πάνω από την έκδοση ήταν το ενδιαφέρον ε, και 125 μονάδες βάσης διαφορά είχαμε 1,2% δηλαδή υπέρ της απόδοσης των δημοσίων ομολόγων σημαντική ε, μείωση σε σχέση με την τιμολόγηση προηγουμένων συναλλαγών στην υπεράκτια μεταφορά Ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών και εξασφάλισε καλύτερες συνθήκες για τη μακροπρόθεσμη επένδυση σε έργα υποδομής. Όπως μας είπε ο κύριος Καζόνη, ε, επίκειται χρηματοοικονομικό κλείσιμο άλλων συναλλαγών, παραδείγματος χάρη στον τομέα μεταφορών, ε, μεταφορών συγγνώμη, θα έχουμε τον ε, αυτοκινητόδρομο Α11 στο Βέλγιο. Αυτή την εβδομάδα θα γίνει με επίσημο, επίσημη εκδήλωση το Σαββατοκύριακο. Ε, πρόκειται για πρόγραμμα εκμετάλλευσης ανεκμετάλλευτης ζώνης, Greenfield Project, και αυτά τα προγράμματα εν μέρη είχαν σχεδιαστεί, θα αρχίσει η κατασκευή με την επίσημη εκδήλωση, θα βγάλουν το πρώτο φτιάρι στην άσφαλτο, αρχίσουν να σκάβουν δηλαδή. Ε, χρηματοδότηση για τέτοιου είδους ε, προγράμματα ανεκμετάλλευτων ζωνών είναι μια θετική εξέλιξη. Ε, πέραν αυτού όμως τα ομόλογα θα εκδοθούν επί τη βάση των αναγκών του προγράμματος, δηλαδή επί τη βάση των κατασκευαστικών αναγκών του προγράμματος. Έτσι έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση και ξαναλέω είναι προς όφελος των, της αναθέτουσας αρχής και του φορέ ε, εκμετάλλευσης ε, του έργου. Ε, παραλλήλου υπάρχει η διαδικασία εξέτασης άλλων εναλλακτικών λύσεων από τον τραπεζικό τομέα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τελικά προέκριναν την έκδοση ομολόγου, ομολόγων έργων λόγω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθήκων. Προχωρώ και βάσει του χρονοδιαγράμματος της πιλωτικής φάσης έχουμε εντοπίσει διάφορα ε, προγράμματα υψηλής δυναμικότητας, 1,2 ε, δις ε, είναι ο σχεδιαζόμενος προϋπολογισμός. Φυσικά θα προσθεθούν κατά πάσα πιθανότητα και νέα προγράμματα. Ο ορίζοντας για την πιλωτική φάση είναι μέχρι τα τέλη του 2014 να εγκριθούν αυτά τα προγράμματα. Η ΕΤΕΠ ε, βεβαίως λαμβάνει υπόψη την απόφαση για την ε, διευκόλυνση διδάση στην Ευρώπη ε, βάσει της οποίας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις μέσα στο 2014-2015 για να μην υπάρξει κενό στη χρηματοδότηση. 1,200 εκατομμύρια ε, πιστοτικής ενίσχυσης λοιπόν αυτό οδηγεί σε υψηλότερο όγκο χρηματοδοτικό δηλαδή σε σχέση με την υποστήριξη του χρέους που ε, καθιστά δυνατό αυτό το ποσό και ε, το κόστος που υποστηρίζουν οι ίδιοι οι επενδυτές ε, βλέπετε ότι η πιστοτική ενίσχυση είναι μικρό κομμάτι ε, της συνολικής χρηματοδότησης του έργου. Ας δούμε τα, το feedback, τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τη μέχρι τούδε εμπειρία η πρωτοβουλία δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το 2012 τον Νοέμβρη υπογράψαμε τις συμφωνίες, ε, είδαμε την εμπειρία του 2013, τώρα έχουμε φτάσει στο 2014 και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό στην αγορά για, σε σχέση με τη ζήτηση των θεσμικών επενδυτών για ε, μακροχρόνια χρηματοδότηση υποδομής. μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τα ομόλογα έργων, αυτό απηχείται ε, συγγνώμη, αυτό μπορεί να αποδοθεί στους ευνοϊκούς ε, χρηματοοικονομικούς ε, όρους, κυρίως για τους δημόσιες αρχές που δρομολογούν και εκμεταλλεύονται τα έργα. Στις αγορές Υπάρχουν προγράμματα που δεν είναι επιλέξιμα για αυτή την πρωτοβουλία και χρησιμοποιήθηκε η ιδιωτική επένδυση σε διμερή βάση. Χρηματοδοτήθηκαν δηλαδή από διεθνού επενδυτέ. Αλλά τι γίνεται με την πρωτοβουλία ομολόγων έργου. Ε, οι δύο εκδόσεις ομολόγων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ε, το πρόγραμμα Κάστορ ε, και Κάφπορ για την μεταφορέα ενέργειας από το υπεράκτιο πάρκο ε, έχουν ε, υποστηρίξει την πρωτοβουλία. Το 2014 ε, δείχνει αυξημένο δυναμικό με αυτό το πρόγραμμα ανεκμετάλλευτης ζώνης στο οποίο αναφέρθηκα στο Βέλγιο. Υπάρχει όμως, υπάρχουν δυνατότητες στην Ιρλανδία, στην Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Άρα θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση ως προς τις χώρες και το είδος προγραμμάτων. 5 ως εφτά προγράμματα ε, θα έχουμε εν τέλει. Αυτός ήταν το στόχος ε, της πιλωτικής φάσης. Και όπως σας είπα, είχε καταλητική σημασία η πρωτοβουλία διότι εστιάζει το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών στη στήριξη ε, της χρηματοδότησης υποδομής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕΠ νομίζω συνέβαλαν ε, σε αυτό επίσης, σε μεγάλο βαθμό. Ε, τώρα, για το μέλλον, για τα προγράμματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, βασικός στόχος είναι να δούμε οι δημόσιε αρχέ, πόσα προγράμματα θα δρομολογήσουν και αυτό φυσικά συνδέεται με ε, τη ε, διαθεσιμότητα πόρων σε εθνικό επίπεδο ε, και θα δούμε ποια προγράμματα κολεύουν να φτάσουν στο δημοσιονομικό κλείσιμο Πάντως το 2013 με τα αποτελέσματα που είχαμε είδαμε αποδείξεις ε, ότι όπως το Βέλγιο για τον αυτοκινητόδρομο ε, Α11 καταφέραμε να βελτιώσουμε την περαιτέρω τις ε, χρηματοδοτικές συνθήκες για τους δημιουργικούς επενδυτές, δηλαδή ανταποκρίνονται αν θέλετε οι επενδυτές σε αυτά τα προγράμματα. Φυσικά για την πιστοτική ενίσχυση θα το ενδιαφέρον μας στα προγράμματα που έχουν προσθέμενη αξία σε σχέση με τη χρήση αυτού του εργαλείου ενδιαφερόμαστε κυρίως για χώρε και προγράμματα όπου πραγματικά ε, η πιστοτική ενίσχυση μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ε, ε, εντείνει το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών σε σημαντικό βαθμό. Φυσικά το σημαντικό είναι οι αποφάσεις των οργανισμών αξιολόγησης επιστοληπτικής ικανότητας. Θα δούμε λοιπόν πώς η πιστοτική ενίσχυση ε, εκλαμβάνεται από αυτούς τους οργανισμούς. Ε, για το πρόγραμμα Α11 η βαθμολόγηση θα περάσει από τη χαμηλή βαθμίδα, ε, δηλαδή τριπλό β με αρνητικό πρόσημο. και φτάνει στο α μείον, νομίζω ότι αυτός ήταν ε, μεταξύ άλλων ο στόχος ε, του προγράμματος ε, της επιστοτικής ενίσχυσης. Εν τέλει να πω κάποια πράγματα για τη μελλοντική πορεία και το πώς θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας σε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν. Οι ανεκμετάλλευτες ζώνες ε, πιστεύω ότι είναι στον πυρήνα της πρωτοβουλίας και η πρώτη συναλλαγή που θα γίνει για τέτοια ζώνη έχει ισχυρό δυναμικό για περαιτέρω συναλλαγές ε, για το 2014 και ε, για αργότερα οι θεσμικοί επενδυτέ θα δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι μπορούν να ανταποκριθούν στι ανάγκε των προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία έχει ισχυρό ρόλο στον τομέα επίση τη τυποποίηση. Δηλαδή ενδιαφέρει του θεσμικού επενδυτέ στην ε, υποδομή το θέμα τη τυποποίηση, ε, Δηλαδή αυτό που επιζητούν είναι κοινά χαρακτηριστικά σε αυτά τα προγράμματα. Δεν θέλουν να υπάρχουν σημαντικέ ε, διαφορέ ανάμεσα στα προγράμματα θέλουν να υπάρχουν ε, κοινά σημεία, αυτό που τραβάει περισσότερο το ενδιαφέρον τους ε, στη συνέχεια προγράμματα θα υπάρξουν στη Νότια Ευρώπη. Σας υπαρχήσαμε από την Ισπανία, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πιο πλούσιο μίξ ε, χωρών, αλλά και την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου προβλέπονται ήδη κάποια προγράμματα. Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε επίσης το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας, ε, όπως είπαμε και σε αρχικές, αρχικά στάδια των συζητήσεων, θα βασιστούμε στα προγράμματα που ε, στρέφονται στην αγορά, διότι αυτό το εργαλείο ε, είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες της αγοράς. Όταν είναι όριμα τα προγράμματα και φτάσουν στο σημείο να ανοιχτούν στις αγορές, τότε θα επέμβουμε εμείς σε σχέση με την ε, χρηματοδοτική διευκόλυνση συνέντα στην Ευρώπη, η ΕΤΕΠ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να δώσει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιες αρχές για την ίδια την πρωτοβουλία. Ε, αυτό είναι ένα σημείο που επεξεργαζόμαστε ήδη στα πλαίσια του Συνδέοντα στην Ευρώπη και οι αναθέτουσε αρχέ επίση θα θέλαμε να δείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τι νέε δυνατότητε των θεσμικών επενδυτών, ούτω ώστε να δουν ε, οι διαδικασίε ανάθεση με ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν πιο εύκαμπτε και να προσαρμοστούν περισσότερο στι ανάγκε των θεσμικών επενδυτών. Ευχαριστώ. Και, και εγώ ευχαριστώ κύριε Μέρφη. Έχω διάφορους που έχουν ζητήσει το λόγο μεταξύ αυτών, Λίχτεμπεργκερ, άλλοι. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές. Θα ήθελα να κάνω ερωτήσει για τον τρόπο λειτουργίας για τα δικτύα ε, συνδέω στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι βαθμό έχετε κάνει όλη την προπαρασκευή για να λειτουργούν στα πλαίσια της χρηματοδότησης. Τι συνεργασία έχετε με αυτούς που έχουν αναλάβει το πρόγραμμα. Δεύτερον, ερωτήσεις για το σε τι θα χρησιμεύσουν, πώς θα αξιοποιηθούν αυτά, πόσο κοστίζει για κάποιον ο οποίος θα προωθεί η χρήση τους. Καταλαβαίνω ότι δεν το κάνουν για κοινοφελείς ε, αφιλοκερδός. Θέλω να μάθω λοιπόν τι κόστος έχουν αυτά. Και δεύτερον, η ΕΤΕΠ συνδέει αυτά τα ομόλογα έργου ως πακέτο μαζί με άλλες μορφές χρηματοδότησης μπορούν να προσφερθούν και αυτόνομα. Αυτές είναι οι τρεις απλές νομίζω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάσνα. θα με ενδιέφερε να καταλάβω γιατί δεν υπήρξε σωστή πιλωτική φάση. Αυτή είναι τώρα η πολιτική φάση. Διότι νομίζω ότι είχαν δεσμευτεί πιστώσεις ε, να γίνει πρώτα το 12 και το 13 μια πιλωτική φάση. Υπήρχαν βέβαια μεγάλες προσδοκίες για αυτό το πρόγραμμα ότι θα υπήρχε μεγάλη ε, μόχλευση, δηλαδή δυνατότητα συγχρηματοδότηση. Συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Αυτή είναι τώρα η πιλωτική ή η ουσιώδης φάση. Και επίσης, ως ε, ΕΤΕΠ, τι επίπεδο μόχλευσης θέλετε να επιτύχετε ή στοχεύετε να επιτύχετε. Όλοι Ρεν είπε ότι θα μπορούσε η μόχλευση να φτάσει στο επί 20 Θαυμάσιο θα ήταν, αλλά ρεαλιστικά, τι μόχλευση έχετε επιτύχει ήδη για αυτά τα προγράμματα, τα ομόλογα έργου. Και τρίτη ερώτηση. Τι θα γίνει με την Ανατολική Ευρώπη. Εκεί υπάρχει μεγάλη ανάγκη υποδομών, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη. Έχει να κάνει με το ότι η συγχρηματοδότηση δεν είναι δυνατή, δεν έχουν υπάρξει αιτήσει ε, για προγράμματα. Βεβαίω είμαι από τη Δυτική Ευρώπη, αλλά με ενδιαφέρει ολόκληρη η Ευρώπη. Ο κύριο Κράμερ Βεβαίως αυτά τα ομόλογα ε, τα φτιάχνουμε για να βρούμε χρήματα που δεν έχουμε. Στην παρουσίασή σας είπατε 8 ή 10 φορές ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών. Και είπατε βεβαίως οι επενδυτές δεν θέλουν ε, οποιοδήποτε αλλά συγκεκριμένα προγράμματα. Φυσικά υπάρχουν διάφορα προγράμματα που αντιμετωπίζονται θετικά γιατί έχει κανείς ε, πολύ κέρδος και άλλα που τα αντιμετωπίζουν αρνητικά στην Ελβετία είχε γίνει μια συζήτηση για ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω συγχρηματοδότηση από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και είχε γίνει αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν καλά προγράμματα από τα οποία κερδίζουμε. Δεν θέλουμε όμω αυτά να τα δώσουμε στον κλάδο, θα τα κάνουμε μόνοι μα. Και αυτά τα οποία είναι αδύνατα, ο ιδιωτικό τομέα δεν τα παίρνει. Έτσι είναι τα πράγματα. Ε, περί αυτού πρόκειται. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα αλλά ε, τα πολλά χρήματα που έχουμε για τις μεταφορές δεν τα αξιοποιούμε σωστά στη Γερμανία. Από το 1994 προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τους σιδηροδρόμους. 20 χρόνια δηλαδή προσπαθούμε. Σε αυτά τα 20 χρόνια όχι μόνο έχουν αυξηθεί 15 φορές οι τιμές, αλλά επενδύθηκαν 80 δις και ο απολογισμός είναι ότι για τις ε, μεταφορές μεγάλων αποστάσεων έχουμε λιγότερους επιβάτες ε, από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Αν είχαμε προσθέσει 20 δισεκατομμύρια τέτοιων ε, ομολόγων έργου θα είχε βελτιωθεί τόσο πολύ κατάσταση. Ποιος ενδιαφέρεται. Εάν είναι πιο εύκολη η χρηματοδότηση δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερα τα προγράμματα. Και εδώ και 30 χρόνια μας λένε ότι για τα συγχρηματοδοτούμενα από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αυτή είναι η λύση. Αλλά το θέμα είναι, και αυτό μας λένε οι επενδυτές, ότι αν άξιζε, αν θα είχαμε αρκετό κέρδος, τότε θα το κάναμε. Βεβαίω. Κανείς δεν μπορεί να μας πει ποια ήταν η θετική μας εμπειρία μέχρι τέλους από κάποια προγράμματα. Το 2000 είχε οριστεί ένα πρόγραμμα για τη Φιλανδία που θα έπρεπε να τελειώσει μέχρι τότε και ήταν όλα καθορισμένα και το κόστος και έχει κοστίσει δύο φορές παραπάνω. Μπορώ να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί. Και ρώτησε και η Γκεζίνε Μάισνερ, ποια είναι τα πιλωτικά προγράμματα. Μπορείτε να μας δείξετε ένα πρόγραμμα όπου έγινε σωστή πρόγνωση, σωστή εφαρμογή και πως το τέλος είχαμε το αποτέλεσμα που αναμέναμε. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε αν μπορούμε να επεκτείνουμε. Βεβαίως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά από την πείρα μου με την ιδιωτική χρηματοδότηση είμαι ιδιαίτερος σκεπτικιστής. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, προβλεπόταν πιλωτική φάση διετής με περιορισμένη χρηματοδότηση 250 εκατομμύρια ετησίως. Αν ε, βλέπω εδώ το κανονιστικό πλαίσιο, δεν έχουμε καθορίσει τι θα γίνει στο τέλος της πιλωτικής αυτής φάσης. Μετά την πιλωτική φάση υπάρχει μια αποτίμηση. Πόσο θα μας πάρει αυτή η αποτίμηση 3, 6, 12 μήνες. Και κατά τη φάση αποτίμησης υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν τέτοια ομόλογα έργου ή απλώς περιμένουμε το αποτέλεσμα της αποτίμησης. Δηλαδή για δύο χρόνια έχουμε 250 εκατομμύρια. Μετά τι γίνεται. Όταν τελειώσει η αποτίμηση έχει μια δουλειά η αποτίμηση. Όταν τελειώσει η πιλωτική φάση μέχρι να τελειώσει μετά η αποτίμηση δεν υπάρχουν πιστώσεις. Δεύτερη ερώτηση. Δυο φορές ήδη άκουσα πώς πάνε τα προγράμματα και δεν είδα τίποτα που να μην αφορά τις οδικές μεταφορές. Θα γίνει κάτι γι' αυτό. Ιδιαίτερα για τους υδροδρόμους ή τις εσωτερικές ε, υδάτινες οδούς. Τρίτη παρατήρηση. Το ότι συνεργάζεστε με τις εγγυήσεις των ε, δανείων για τις διευρωπαϊκές μεταφορές Αυτό έχει ήδη προχωρήσει. Υπάρχει αυτή η συνεργασία. Είναι δομημένη για να υπάρχουν προγράμματα, ομόλογα έργου γι' αυτό. Λίχτενμπεργκ. Ευχαριστώ για την εκθεσή σας. Διαπιστώνω ότι είναι πολιτική υποδομών, όχι πολιτική. Είναι πολιτική δημοσίων έργων, όχι μεταφορών. Έχουμε μιλήσει πολύ συχνά για το πώς πρέπει να αποσυνδέσουμε τα θέματα της, ε, των μεταφορών από την ε, από την ε, έκκληση περισσότερου διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ έχουμε αποσυνδέσει πλήρως τα δημόσια έργα από τις μεταφορές και αυτό οξύνεται ακόμη περισσότερο διότι οι ιδιωτικοί επενδυτές πρώτα απ' όλα ενδιαφέρονται για μικρότερα, πιο διαφανή προγράμματα όπου βέβαια υπάρχει κίνδυνος τελικά ε, τον κίνδυνο να τον φέρουν οι φορολογούμενοι και τα κέρδη ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η τάση κατακαιρματισμού που έχουμε στην Ευρώπη για τις μεταφορές αυξάνεται. Θα ήθελα να μάθω σε τι βαθμό ε, αντιμετωπίζεται συνολικά την πολιτική των μεταφορών όπως ακριβώς τη θέτουμε εμείς ως Κοινοβούλιο, με γενικούς στόχους, από τη Λευκή Βίβλο. Αυτά τα λαμβάνετε υπόψη στη λήψη αποφάσεών σας. Είναι... Γίνεται αυτό ή απλώς βλέπετε, αν αυτός κάτι θέλει να φτιάξει, να το χρηματοδοτήσουμε. Θα ήθελα να μάθω αν αυτά που αποφασίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις για τις επενδύσεις σας, στις κρίσεις σας για ενδεχόμενες επενδύσεις. Λαμβάνονται καθόλου υπόψη παίζουν κανένα ρόλο ή είναι εντελώς αποσυνδεδεμένα. Δεύτερον, είναι σαφές ότι στον τομέα των δημοσίων έργων υπάρχει ψηλό επίπεδο διαφθοράς. Αυτό είναι γνωστό. Γενικώ γνωστός. Γνωστό. Έχουν γίνει πολλές ε, επιστημονικές μελέτες που το έχουν ε, τεκμηριώσει. Όταν λέμε λοιπόν να μην υπάρχει κίνδυνος για τους επενδυτές, βεβαίως τους αρέσει αυτό, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουμε ειδικέ προβλέψεις για να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Διότι διαπιστώνουμε ότι στον τομέα αυτό οι υπερβάσεις ε, του προβλεπόμενου κόστους είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση έγινε μια μελέτη γενικά στην Ευρώπη και διαπιστώσαμε ότι οι υπερβάσεις κόστους για τις υποδομές μεταφορών είναι μεταξύ 60 και 200%. Δηλαδή γίνεται αρχική ε, μειωμένη πρόβλεψη και μετά αυξάνεται πολύ το κόστος κατά την κατασκευή. Είναι πολύ εκτεταμένο αυτό το φαινόμενο. Τι κάνετε λοιπόν ε, για να έχετε προβλέψεις για το τι βάρος ε, μεταφορών θα υπάρχει, δηλαδή τι βάρος κυκλοφορίας θα υπάρχει. Ποιος το αποφασίζει αυτό, το δίνεται σε ιδιωτικούς ε, φορείς ανεξάρτητους ή σας το κάνουν τις ε, προβλέψεις για το τι κυκλοφορία θα υπάρχει μετά θα τις κάνουν αυτοί που αναλαμβάνουν το έργο. Υπάρχουν ορισμένα εντυπωσιακά παραδείγματα. Τρίτο ερώτημα για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Στη Βόρεια Ιταλία άκουσα ότι ο περιφερειακός του Μιλάνου θα χρηματοδοτηθεί έτσι. Δηλαδή για άλλη μια φορά ε, ευνοούμε για όλα τα ίδια μεταφορών και ατόμων και εμπορευμάτων και παραδόσεων όλα αυτά ευνοούμε και πάλι τις οδικές μεταφορές έναντι των σιδηροδρόμων. Άρα πώς εξυπηρετούμε τους στόχους του συνδέοντα στην Ευρώπη. Γιατί θα δώσουμε πιστώσεις και από αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν θα μπορούσαν να υπάρξουν ομόλογα έργου για αυτό το έργο. Νομίζω πως είναι παρακινδυνευμένο οι υποδομές των μεταφορών διότι διαπιστώνει επίσης είναι λογικό να ξεκινάμε με μικρότερα έργα όπου είναι ε, αρκετά πιο εύκολο να δούμε τις επιπτώσεις παρά να επιλέξουμε ε, μεγάλης έκτασης υποδομές που βεβαίως παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη βιωσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τέλος ε, θα θέσω ερωτήσεις εγώ. Κύριε Κασόνη, μιλήσατε για ηθικές ασφαλιστικές εταιρείες, μα υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το είχα καταλάβει μέχρι στιγμής. Στις μονογραμμικές... Ναι, ναι, μονογραμμικές... Είπα, δεν είπα moral, είπα μόνο line μονογραμμικές και όχι ηθικές. Πάντως κάτι που ήθελα σοβαρά να πω, είναι κάτι που είπαν και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι. Ε, βλέπω ως ιδιώτες επενδυτές και τον αυτοκινητόδρομο Α11 ε, και να σκέφτονται να ωραία μια καλή ευκαιρία και τα λοιπά, να επενδύσουμε, θα βγάλουμε τα λεφτά μας για την ενέργεια, ναι το καταλαβαίνω. Αλλά το θέμα για μας εδώ στις μεταφορές είναι πόσες φορές θα έχετε ε, παραπάνω εγγραφή ε, άμα ας πούμε πρέπει να ανανεωθούν οι σειρμοί σε ένα παλιό δίκτυο σιδηροδρόμων. Πόσες φορές θα έχετε υπερβολική παραπανήσια εγγραφή άμα θα πρέπει να ανανεωθεί ε, ένα παμπάλαιο τούνελ ας πούμε στις Άλπεις. Άμα δούμε τι γίνεται στη δική μου τη χώρα, η Βρετανία διαρκώς σκάβει τούνελ. Σε λίγο θα μπαίνουμε σε ένα τούνελ από το Λονδίνο μέχρι το Μάντσεστερ, αλλά το θέμα είναι ότι τα, οι σύραγγες αυτές είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Το θέμα που θέλω να πω είναι Πόσες φορές νομίζετε πως θα έχετε τόσο μεγάλη εγγραφή σε αυτά τα ομόλογα έργο, γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτά τα ομόλογα έργο ε, υπάρχουν για να μπορέσουν να υπάρξουν επενδύσεις όταν η ιδιωτική αγορά δεν έχει ε, παρουσιάσει, το, ε, δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ποια είναι τα έργα, πού είναι τα πιλωτικά έργα για αυτά τα περιθωριακά έργα. Ας πούμε όταν αρχίσαμε να μιλάμε για ε, υπηρεσίες βαθμολόγησης ε, ή αξιολόγησης, ε, ποιος, ποιος τις αξιολογεί αυτές, σε ποιον είναι αυτές οι υπόλογες λέγαμε τότε που το συζητάγαμε αυτά τα θέματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να ξέρω ποια είναι αυτά τα περιθωριακά project, τα προγράμματα, άμα επιτρέπετε να τα ονομάσω έτσι, που βρίσκονται αυτά. Και ιδιαίτερα αυτά που ε, περιλαμβάνουν σιδηροδρόμους, σύνδεση με λιμένες, όπου οι ιδιώτες επενδυτές δεν βλέπουν να ανάβουν λαμπάκια με, ευρώ μόλις σκέφτονται ένα τέτοιο project. Ε, κύριε Κασόνη, θα πάρετε εσείς πρώτα το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένε και μετά ο κύριος Μέρφη θα απαντήσει στις υπόλοιπες και αν φυσικά αν έχετε άλλες ερωτήσεις θα επανέλθουμε. Πού βρισκόμαστε τώρα. Τώρα βρισκόμαστε στην πιλωτική φάση από δημοσιονομική άποψη που έτρεχε από το 2012 μέχρι το 2013 η έγκριση των προγραμμάτων ε, θα γίνει μέχρι τις 2014 και η φάση εφαρμογής μέχρι το 2015-16. Ε, στην διευκόλυνση για την ε, συνδέοντα στην Ευρώπη, Ευτυχώς προβλέπεται η συνέχιση της πρωτοβουλίας με προϋπολογισμό που μπορεί να ε, δοθεί στη διάρκεια του 2014 και του 2015 ώστε να μην υπάρξει πάυση όταν, ε, όσον αφορά την μόχλευση θα γίνει πλήρης αξιολόγηση το 2015, αλλά το γεγονός ότι έχουμε προπολογισμό για το 2014 και το 2015, αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης. Όταν αφορά την μόχλευση, όταν λέμε 15 με 20, ο υπολογισμός μας ήταν ότι αυτό, αυτή είναι η μόχλευση του, του κοινοτικού προπολογισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης. Τώρα, όταν δούμε τις ρυθμίσεις ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και την ΕΤΕΠ, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός αναλαμβάνει την πρώτη ζημία που φτάνει μέχρι το 30% ενώ η χρηματοδότηση της ΕΤΕΠ είναι πάνω από τρεις φορές ο προϋπολογισμός της Ένωσης. Έπειτα, εφόσον η ΕΤΕΠ μπορεί να αναλάβει μόνο το 20%, μόνο το 20% της έκδοσης των ε, ομολόγων σημαίνει πως είναι πενταπλή η μόχλευση ανάμεσα στην ΕΤΕΠ και τον τελικό εκδότη του ομολόγου. Δηλαδή 15 με 20 φορές τον προϋπολογισμό της Ένωσης φτάνουμε έτσι. Ελπίζω πως έτσι σας αποσαφήνισα το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα, από τη δική μας ε, άποψη, ε, εικόνα μάλλον, προοπτική, ε, νομίζω πως σας δείξαμε ότι η αγορά των ομολόγων εξυφανίστη. Ήταν ένα μέσο χρηματοδότηση μέχρι κάποια στιγμή και μετά εξαφανίστηκε από την αγορά για κάποια χρόνια. Όταν μαζί με την ΕΤΕ προσπαθήσαμε να προτείνουμε αυτή την νέα ιδέα, θελήσαμε να αναζωογονήσουμε την αγορά και να διευκολύνουμε την ε, έκδοση των ομολόγων από τους θεσμικούς επενδυτές. Να ξαναδημιουργήσουμε στην ουσία μια αγορά ομολόγων και από την ανταπόκριση της αγοράς και εν γέννη ως γενική εξέλιξη νομίζω πως ήταν θετική η αντίδραση γιατί η αγορά όντως έχει ξεκινήσει και πάλι. Όταν θα περάσουμε στην επόμενη φάση, μετά την πιλωτική, ε, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό και η ΕΤΕΠΑ θα σας το πει και εκείνη, ότι αυτό δεν είναι ανοιχτό μόνο για τις νέες χώρες όπου όντως οι υποδομές θα πρέπει να βελτιωθούν ε, ε, και πιθανά σε νέους τομείς. Έχουμε μια ιδέα επίσης στην Κομισιό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, ώστε αυτή η λύση από τη στιγμή που θα έχει αποδείξει την αξία της να υπάρχει και για την ε, στις βιώσιμες μεταφορές αλλά και για άλλους τομείς που είναι πιο στην, στο περιθώριο θα λέγαμε. Αλλά για να επανέλθουμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως, πιστεύω πως ό,τι και αν κάνουμε, ε, χρηματοδότηση έργου ή ομόλογα έργου, ε, για μας το σημαντικό και για το Κοινοβούλιο νομίζω το ίδιο, γιατί είμαστε ε, στο ίδιο μήκος κύματος, αυτό είναι καλά ε, προγράμματα, καλά έργα για το κοινό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τα ομόλογα έργο είναι να βοηθήσουμε ώστε να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο οικονομικό και πιο φθηνό για τον ε, κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέγα θέμα ρευστότητας, αλλά μάλλον έλλειψη καλών ε, σχεδίων. Και εδώ πρέπει να ενεργήσουμε μέσω τη διευκόλυνση για τη διασύνδεση, τη, διευκόλυνση τη συνέοντα στην Ευρώπη. Πώ θα μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε καλά σχέδια που να έρθουν στην αγορά και έπειτα να χρησιμοποιήσουμε τεχνικέ και εργαλεία όπως τα ομόλογα έργου για να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε. Αλλά δεν είναι, γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ομόλογα έργου ξαφνικά θα εμφανιστούν και καλά σχέδια ε, έργα. Ε, θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει ένα καλό πρόγραμμα, αξιοπιστία, διαφάνεια και μέσω του ομολόγου έργου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους όρους της πίστοσης και να ελκύσουμε την αντίδραση των επενδυτών. Τώρα, αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι το ομόλογο έργο συνδέεται αυστηρά με την προηγούμενο κανονισμό για την πιλωτική φάση και την διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη για την επόμενη φάση. Τα προγράμματα δηλαδή που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς. Η ΕΤΕΠ θα πει το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε άλλους τομείς μέσω της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη, γιατί ελπίζουμε πως αυτό θα είναι στην ευρωπη γιατι ελπιζουμε πως αυτο θα ειναι εφικτο Αυτό που είναι όμως σημαντικό πέρα από αυτό το τομέα είναι η ικανότητα της ΕΤΕΠ και το λέω αυτό εξ ονόματος της Κομισιόν, η ικανότητα της ΕΤΕΠ να αξιολογεί τα προγράμματα ε, ενδελεχώς έχουν πολύ σημαντικές ε, προδιαγραφές ας πούμε για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων ε, και για ε, τον έλεγχο της συμμόρφωσης ας πούμε με τις οδηγίες του περιβάλλοντος είναι πάρα πάρα πολύ ενδελεχής όσον αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προχρωμάτων, ώστε να αποφευθεί διαφθορά και να μην μπούμε σε, ε, νερά. Θα ζητήσω τώρα από τον ε, και να εστιάσει περισσότερο στο θέμα των όρων χρηματοδότησης και στα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις προβλέψεις για το φόρτο της κυκλοφορίας και ποια είναι τα προγράμματα που ε, προετοιμάζονται. Λοιπόν, να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά για τις ε, συμβουλές που λαμβάνουμε και πώς μπορούν οι εταιρείες συμβούλων και οι υπηρεσίες που παρέχουν να μας βοηθήσουν. Υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες, υπάρχει το κέντρο γνώσης για τις πρωτοβουλίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προσπαθεί να καταστήσει γνωστές εθνικές αρχές τις βέλτιστες πρακτικές στην πολιτική όπως ανάφερα δημοσίων προμηθειών ούτως ώστε να είναι όσο πιο προσαρμοσμένη και ευλίγιστη γίνεται και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συμμεριζόμεθα εμπειρίες με τις εθνικές αρχές, πώς να βοηθήσουμε τα προγράμματα τώρα, πώς να ενισχύσουμε τα καλύτερα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα ε, δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται με ομόλογα. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλο τα, όλα τα προγράμματα. Χρηματοδοτούμε γενικά προγράμματα του δημόσιου, του δημόσιου τομέα και είναι σημαντικό τμήμα αυτό της δουλειάς μας και στα προγράμματα όπου υπάρχει ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση οπωσδήποτε συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα γίνουν αυτά τα προγράμματα ιδιαίτερα εκεί που χρειάζεται να βοηθήσουμε τις δημόσιες αρχές. Τώρα το κόστος της πρωτοβουλίας, τι δηλαδή χρεώνει η ΕΤΕΠ ε, είναι το λεγόμενο κεφαλαιακό κόστος, το κόστος του κινδύνου. Δηλαδή κάνουμε τον υπολογισμό. Δηλαδή προσπαθούμε να ε, βγάλουμε το κόστος μας. Δεν επιδιώκουμε να έχουμε υψηλού επίπεδου κέρδου σαν να ήμασταν ιδιωτικό τομέα. Για την πιλωτική φάση τώρα στοχεύουμε στην αξιολόγηση που θα γίνει το 2015 που θα βασιστεί στο τι θα γίνει το 13 και 14. ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε σωστά τι επετεύχθη. Να δούμε δηλαδή αναλυτικά τα προγράμματα, να δούμε τι ρόλο καταλήτη έπαιξε αυτό το μέσο, πώς τα πήγαν τα προγράμματα. Τι μόχλευση τώρα. Θα έλεγα ότι η φύση των ε, χρηματοδοτήσεων, δηλαδή 200 για τις μεταφορές, 200 για ευρυζωνική τηλεπικοινωνία και 200 εκατομμύρια για την ενέργεια. Τα πρώτα δύο προγράμματα, το Κάστορ και το δεύτερο, διαπιστώσαμε ότι είχαν μία χρηματοδότηση 1,8 ε, δις, ενώ η δική μας χρηματοδότηση ήταν μόνο 10 εκατομμύρια. Υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Βέβαια αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Ε, έχει να κάνει με το ότι είχαμε περιορισμένες δυνατότητε, περιορισμένες πιστώσεις για θέματα ενέργειας σε αυτήν την πιλωτική φάση. Ενδιαφέρον των επενδυτών για καλά προγράμματα. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη προσέγγιση μας, ότι μόνο καλά προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτούμε. Όταν ε, αναλαμβάνουμε συμπληρωματικούς κινδύνους πέραν των συνήθων, αυτό σημαίνει πως θεωρούμε ότι είναι καλά προγράμματα, ποιοτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα προγράμματα ε, πρέπει να γίνονται από τις ε, πλουσιότερες περιοχές, ότι πρέπει να, αλλά ότι πρέπει να είναι καλά δομημένα, και να αντιμετωπίζονται σωστά οι κίνδυνοι. Η λειτουργία τώρα της ΕΤΕΠ αφορά όλη την Ένωση, όλες τις περιφέρειές της. Οπότε αυτό είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε πάντα. Πάντα θέλουμε να υπάρχει σωστή διαχείριση και σωστή δομή. Τώρα, ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, μέσων μεταφορών. Ε, ας πούμε να σας πω για το περιφερειακό του Μπορτό τα τελευταία δύο χρόνια το, την λιμενική είσοδο του Λονδίνου επίσης Τώρα, για την πιλωτική φάση των ομολόγων έργου, πρόκειται για έργα τα οποία είναι σε υψηλό επίπεδο οριμότητα και μπορούν να εγκριθούν από την ΕΤΕΠ μέσα στο 2013 14 ανάλογα με το ποια έργα τώρα οριμάζουν σε αυτή τη φάση. Και είναι σωστό να πει κανεί ότι ιδιαίτερα στο σιδηροδρομικό τομέα και τη χρήση ιδιωτική χρηματοδότηση δεν υπήρξαν πολλά προγράμματα σε αυτή τη φάση τη χρονική. Σαφώς υπάρχουν σημαντικά προγράμματα για το μέλλον, αλλά το συγκεκριμένο τομέα δεν είναι πολλά. Η ΕΤΕΠ, ωστόσο, είναι πρόθυμη να στηρίξει ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω των ομολόγων έργου στον σιδηροδρομικό τομέα, αλλά και στον τομέα των εσωτερικών πλωτών οδών. Και αυτό είναι κάτι που το οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ε, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές για να εντοπίσουμε ε, δυνητικά ε, προγράμματα ή έργα. Όσον αφορά την αξιολόγηση που θα γίνει το 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ε, το πώς θα το διαχειριστεί η ΕΤΕΠ ε, για τα κονδύλια δηλαδή που θα χορηγηθούν το 2014 και 2015 και σε ποια φάση θα υπάρχουν τα κονδύλια από το 2015 η συμφωνία ΣΕΦ προβλέπει την επιπλέον χρηματοδότηση για το 2014-2015, επιπλέον 230 εκατομμύρια, οπότε σε κάποιο βαθμό υπάρχει συγχρονισμός. Όσον αφορά όμως τους όρους δέσμευσης ε, υπό το ΣΕΦ για οτιδήποτε πέρα από το 230 εκατομμύρια, αυτό θα εξαρτηθεί από την αναθεώρηση που θα γίνει το 2015 και θα είναι και το αντικείμενο της έκθεσης που θα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα την εγκυοδοσία για τα δάνεια και τα σχετικά, το σχετικό μέσο εξακολουθεί να υπάρχει, μπορούν να εγκριθούν προγράμματα μέχρι τα τέλη του 2014. Το συγκεκριμένο αυτό μέσο εστιάζει στους κινδύνους ε, κυκλοφορίας σας ανέφερα την, την είσοδο στο Λονδίνο και στο το περιφερειακό του Μπορντό ως σχετικά προγράμματα. Σε ολόκληρο όμως στην Ευρώπη στις περισσότερες δικαιοδοσίες γίνονται έργα τα οποία βασίζονται στην, ε, σε, σε πληρωμή κινητικότητας, ε, σε φόρους κυκλοφορίας και όχι σε διόδια ή σε ε, πληρωμή της κυκλοφορίας από συγκεκριμένους δρόμους ή περιφερειακούς. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε. Το ομόλογο έργου συνδυάζεται με την αγορά ομολόγων ενώ το μέσο εγκυοδότησης και δανείων ε, είναι σε βάση, μάλλον λειτουργεί με βάση το τραπεζικό σύστημα. Είναι κάτι το διαφορετικό Γι' αυτό θα κοιτάξουμε πώς στο μέλλον θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο της εγκυδότησης και των δάνειων για να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω των ομολόγων έργου. Τώρα, όσον αφορά και πάλι την επιλογή προγραμμάτων, περιβαλλοντικά και άλλα κριτήρια, ο κ. Καζόνη νομίζω το τόνισε αυτό, πως τα κριτήρια για την πρωτοβουλία ομολόγου έργου ε, αφορά βασικά ε, προγράμματα κατασκευών μεταφορών αλλά και τα ευρυζωνικά. Γίνεται αξιολόγηση και εκτίμηση από πλευρά της ΕΤΕΠ όσον αφορά θέματα όπως η διαφθορά. Φυσικά <laughs> είναι προς αποφυγή. Κατά μια έννοια ε, η υπέρβαση του κόστους και τέτοια θέματα, ένα από τα θέματα τα οποία χαρακτηρίζουν τα προγράμματα PPP ε, είναι υπερβάσεις κόστους αλλά ε, αυτό το προβλέπουμε εμείς και όταν είσαι επενδυτής ή παρέχεις χρηματοδότηση σε ένα πρόγραμμα PPP που βασίζεσαι μόνο και μόνο στο ίδιο το πρόγραμμα για να σου φέρει απόδοση και να σου ξεπληρώσει τα χρήματα που επένδυσες θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές κατευθύνες γραμμές και έλεγχοι ώστε να είμαστε βέβαιοι πως το πρόγραμμα δεν θα παρουσιάζει υπέρβαση κόστους. Τώρα, για τις προβλέψεις για τη φόρτο κυκλοφορίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης PPP, ιδιαίτερα στα προγράμματα που αφορούν την κυκλοφορία και αυτό το εξετάζουμε πολύ προσεκτικά στην ΕΤΕΠ. Έχουμε ένα σύνολο μηχανικών οικονομολόγων που αναλύουν τα προγράμματα Τώρα, σε σχέση με το PPP ή μη PPP. Αυτό είναι ευρύτερο θέμα, ευρύτερη συζήτηση. Η απόφαση ήταν να χρησιμοποιήσουμε ιδιωτική χρηματοδότηση. Η ΕΤΕΠ χρηματοδοτεί πάρα πολλά προγράμματα που δεν υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση. Μάλιστα τα περισσότερα είναι τέτοια και αυτό εξαρτάται από την εθνική οικονομία. Υπάρχουν τώρα ε, δημοσιονομικοί περιορισμοί, περιορισμοί στο δανεισμό. Υπάρχει μια υπόθεση ότι η ιδιωτική συμμετοχή θα είναι σημαντικό μέρος, ε, όχι το κύριο μέρος, αλλά σημαντικό μέρος για τις, ε, για τις χρηματοδοτικές λύσεις του μέλλοντος και για το ομόλογα έργο φαίνεται να είναι ανταγωνιστικά και ελκυστικά ως βάση γιατί παρέχουν βεβαιότητα και στις εθνικές αρχές αλλά και στους ε, ιδιώτες χορηγούς. Τώρα, τα κριτήρια που εφαρμόζει η ΕΤΕΠ αναζητούμε θετική οικονομική απόδοση για τα ε, προγράμματα. Αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο και σε κάποιο βαθμό είναι και ένα ορόσημο για το αν θα αποφασίσουμε για, τον, για την απόφαση που θα λάβουμε αν είναι καλό ή όχι το πρόγραμμα. για τη χρηματοδότηση ε, ε, ε, προγραμμάτων όπου είναι ανύπαρκτη η ιδιωτική αγορά. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι βέβαια να αποφύγουμε ένα κενό χρηματοδότησης όταν μιλάμε για τις σημαντικές ε, ε, επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό μέσω θεσμικών επενδυτών που θέλουν να επενδύσουν σε υποδομές που ωφελούν την κοινωνία των πολιτών. Αλλά όσον αφορά τα προγράμματα, το αν δηλαδή η υπερβολική εγγραφή είναι καλό ε, σημάδι ή κακό σημάδι, από την πλευρά των επενδυτών είναι καλό σημάδι. Αλλά όσον αφορά τα μεμονωμένα, ε, όσον αφορά τα μεμονωμένα τώρα προγράμματα, ε, εξαρτάται από τη χώρα, εξαρτάται από την βαθμολόγησή του, από την αξιολόγησή του, δεν είναι ένα μέσο για αδύναμα προγράμματα, αλλά είναι ένα μέσο που μπορεί να στηρίξει καλά προγράμματα, ώστε να χρηματοδοτηθούν σε κάποια στέρεη βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί αυτά τα προγράμματα από δημοσιονομικής άποψης να είναι κάπως πιο αδύναμα. Τώρα, για τις ε, οργανισμούς ε, αξιολόγησης, είναι σημαντικοί αυτοί οι οργανισμοί για τους επενδυτές, αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο αυτό. Πιστεύουμε πως για τους επενδυτές η συμμετοχή της ΕΤΕΠ είναι ένα σημαντικός παράγοντα όσον αφορά την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις υποδομές γιατί θεωρούν πως έχουν ένα εταίρο που είναι προσιλωμένο στην ολοκλήρωση του έργου ε, ε, μέχρι ότου αυτό αποσβηθεί και ενώ η αξιολόγηση είναι σημαντική, η συμμετοχή ενό δημόσιου οργανισμού είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια για τους επενδυτές. Σας ευχαριστώ. Εντάχει γιατί περιμένουμε και τον Επίτροπο. Ένα λεπτάκι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον αυτοκινητόδρομο το ε, ε, Μιλάνο και γενικότερα για τη Βόρεια Ιταλία σε δρόμους δεν απαντήσατε. Προβλέπετε κάτι γι' αυτό ή όχι. Μα σας είπα για την Ιταλία νωρίτερα. Προβλέπετε, ναι. Εξαρτάται σε ποια χρονική στιγμή θα υλοποιηθεί ποιο πρόγραμμα. Δεν είμαι και ειδικό ε, για τους αυτοκινητοδρόμου, αλλά ο αυτοκινητόδρομος Μπρεμπέμι έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕΠ, από ό,τι ξέρω, ε, και επίσης ε, υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα, περιφερειακός του Μιλάνου, που θα χρηματοδοτηθεί, τώρα δεν ξέρω Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι προτεραιότητες που έχουμε ορίσει σε σχέση με αυτά που εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε το μέλλον της πολιτικής μεταφορών, ε, για τα βέβαια ε, μεταφορών και τις προτεραιότητες. Εφόσον ε, έχω την ιδιότητα του συντονιστή θα πρέπει να στρέφομαι ε, προς την ΕΤΕΠ όταν μιλάμε για χρηματοδότηση υποδομών στους λιμένες και ούτω καθεξής γιατί βάζω στοίχημα τη ζωή μου ότι θα απουσιάζουν οι ιδιωτικοί επενδυτές ε, και, και εκεί κολλάει το πράγμα. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά που θέλουμε να συμβούν στους χώρους που συνιστούν προτεραιότητες για μας. Ε, μας μιλάτε για αυτοκινητοδρόμους, αυτοκινητοδρόμους, αυτοκινητοδρόμους. Για μας δεν είναι προτεραιότητα, τέλος πάντων. αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Ε, κύριοι, σας ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας, για τις απαντήσεις σας. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την Τρίτη, 1η Απριλιά, 9, στην 5G3. Οπότε θα τα δούμε τότε. Και θυμίζω στους συντονιστές ότι θα έρθει στις 11 ο Επίτροπος Κάλλης για να μας κάνει την αναφορά ε, του Συμβουλίου Μεταφορών. Ο Πρόεδρος ευγενικά ευχαριστεί και τους δύο Ευχαριστώ.